Dear colleagues, good morning. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Yes. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν περάσουμε στη ψηφοφορία, θα ήθελα να σας ζητήσω να βάλετε στο μηχάνημα την ε, κάρτα σας, την ηλεκτρονική, για να ξέρουμε πόσοι ε, μπορούν να ψηφίσουν εν μεταξύ. Να σας πω για τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη χθεσινή συνεδρίαση των ε, συντονιστών. Ε, οι οποίες πρέπει να εγκριθούν από την ε, Επιτροπή. Πρώτον, ένα μέλος του ΕΛΚ ε, διορίζεται, ορίζεται ως εισηγητής για τις κοινέ ελάχιστες προδιαγραφές για τις αστικές διαδικασίες. Ε, η κυρία Πεσερόφα είναι η συγκήτρια για τους ευάλωτους ε, ενήλικες. Ε, το ΕΛΚ επίσης έχει αναλάβει την έκθεση πρωτοβουλίας για τις διασυνοριακές αναγνωρίσεις υιοθεσίας. Επίσης για τον περιορισμό των εγώ ίδιος θα είμαι ε, υπεύθυνο για το θέμα του ε, ε, περιορισμού των προβλημάτων με τις αστικές παραβάσεις και επίσης η ECR έχει αναλάβει την γνωμοδότηση για την ε, αναθεώρηση της οδηγίας 2011 κάθετος 16 για την ανταλλαγή πληροφοριών ε, για, το, για τα θέματα ε, φορολόγησης από την ομάδα των, των σοσιαλδημοκρατών, ο κύριος Καρίμ θα αναλάβει το θέμα της επικορικότητας, της επιτροπολογίας και της εκχώρησης των νομοθετικών δραστηριοτήτων ο κύριος Χρυσόγονος, ε, για τις κωδικοποιήσεις η κυρία Χάουταλα. Οι συντονιστές αποφάσισαν ε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση της Reft Club ε, θα προσκληθεί ε, στην Επιτροπή μας ε, τον Ιούλιο και επίσης για την αποστολή στον ΩΣΑ το, στο Παρίσι θα γίνει αλλαγή ημερομηνία για το Σεπτέμβρη του 2015. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις από τη συνεδρίαση των συντονιστών που έλαβε χώρα εχθές. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Προστασία ε, της τεχνολογίας, της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται, εμπορικών απορρίπτων. Θα ήθελα να σας ζητήσω να εισάγετε την κάρτα σας στην ηλεκτρονική στη σχισμή 18 είναι τα μέλη που θα ψηφίσουν. «24 είναι κανονικά, 18, 19, ο κύριος Τζαμπάσκι δεν έχει την κάρτα του». Uh, thank you. We have 24 cards. 24 κάρτες έχουμε πλέον ε, στα μηχανήματα, οπότε εντάξει. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ. Παρακαλώ, ψηλά τα χέρια σας. Κρατήστε τα ψηλά. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία παρήθμων 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 309 υπέρ. Τριακόσια εννέα. Υπέρ. για το άρθρο 11 παράγραφος 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ίμκο 39. Υπέρ. Πάλι για το άρθρο 11. Ίμκο 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 387 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 388 Υπέρ. Κατά. Αποχές να την ελέγξουμε αυτή καλύτερα. σε έναρξη ψηφοφορίας. Είναι πολλοί οι συνάδελφοι που ψηφίζουν. 25 ψήφισαν τώρα. Εντάξει τώρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 310 υπέρ. 310 επαναλαμβάνω υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήτρε 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 92. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήτρε 93 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 94 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήτρε 95 υπέρ, κατά, χέρες εγκρίνεται. 314 υπέρ κατά έλεγχος παρακαλώ εγκρίνεται Ήμκο 41 υπέρ. Ήμκο 41. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήτρε 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τριακόσια δεκαέξι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 317 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Εγκρίνεται. Τροπολογία 321. Υπέρ. Κατά. Καλύτερα να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά και αυτό. Εγκρίνεται. Ήτρε 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 333 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 334 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, απορρίπτεται. Ήμκο 45. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Λοιπόν, ψηφίζουμε την ΙΜΚΟ 45. Σωστά. Δύο ακόμη μένουν να ψηφίσουν. Εγκρίνεται. Τροπολογία 335. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο? Έλεγχος. Ωραία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. ή 3 υπέρ. Κατά. Καλύτερα να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Εγκρίθηκε. Σαραντεπτά. Υπέρ. Κατά. ηλεκτρονικός έλεγχος. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 48. Υπέρ. Κατά. Αποχέρ. Απορρίπτεται. Λοιπόν, αδειολογικη σκέψη 12, α, ήτρε 11, υπερ αδειολογικη Αιτιολογική σκέψη 12α, επαναλαμβάνω, τροπολογία ήτρε 11, υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Ήμκο 7. Υπέρ. Κατά. Καλύτερα να την ελέγξουμε και την ΙΜΚΟ 7. Εγκρίνεται. λογική σκέψη 14, τροπολογία 8, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 69, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 14, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ίμκο 8. Όχι, όχι. Λάθος. Διορθώνει ο πρόεδρος. Ήτρε 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καλύτερα να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Εγκρίνεται. Ήτρε 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Εγκρίνεται. Ήτρε 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη 25α. Τροπολογία 9. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται αλλά καλύτερα να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο εγκρίνεται Αιτιολογική σκέψη 28 Τροπολογία 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήμκο 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του σχεδίου εκθέσης, ηλεκτρονικός υποθέτω. Ωραία. Έναρξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα και το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Μία ακόμη φορά ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Δύο ακόμη συνάδελφοι πρέπει να ψηφίσουν. Πέρα τη ψηφοφορία εγκρίνεται. Και τώρα πρέπει να ψηφίσουμε την απόφαση έναρξης διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Μία ακόμη φορά ηλεκτρονικός. Εγκρίνεται. Σα ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε μία μόνο σοφορία για κάποια θέματα. Uh, may I May ε, θα ήθελα να συγχωρώ την κυρία Λαγκρίπ. Τώρα ε, μία μόνο ψηφοφορία για κάθε θέμα, ηλεκτρονική κάθε ψηφοφορία. Πρώτα το κοινοτικό σήμα. Άρχεται. εγκρίνεται με ευρεία πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στην κυρία Βίξτρομ Κατόπιν νομοθεσία των κρατών μελών για τα σήματα, άρχεται η ψηφοφορία. και πάλι συγχαρητήρια στην κυρία Βίλστραν. Τώρα το πακέτο για τα σήματα και πάλι άρχιτη ψηφοφορία. Ευχαριστώ, εγκρίνεται. Τώρα έχουμε μία ψηφοφορία για Τώρα λοιπόν καταρχάς θα ήθελα ίσως να δώσω το λόγο στην κυρία Βίξτρομ. Δεν χρειάζεται λέει η κυρία Βίξτρομ, ε, μίλησα αρκετά. Άλλη μια φορά σας ευχαριστώ όλους. And we, Ο κύριος Γκρόζα, μήπως από το Συμβούλιο, θα ήθελε να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Σφόποντα. Από πλευρά της Λετωνικής Προεδρίας, ε, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την εργασία για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο. Είμαστε ήδη η πέμπτη Προεδρία του Συμβουλίου που ασχολείται με αυτό το πολιτικά και οικονομικά σημαντικό θέμα. Η, η Ισλανδική, η Λιθουανική και η Ελληνική Προεδρία προσπάθησαν με σκληρή εργασία να επιτύχουν συμβασμό στο Συμβούλιο και η Ιταλική Προεδρία ολοκλήρωσε το συμβασμό στο Συμβούλιο και ξεκίνησε διαπραγματεύσει για μια συμφωνία δεύτερη ανάγνωση. Η Προεδρία μα είχε την τιμή να καταλήξει να βοηθήσει να καταλήξουν αυτές τις διαπραγματεύσεις. Είμαστε πολύ κοντά λοιπόν τώρα να κλείσουμε το θέμα αυτό και η ψηφοφορία σας ε, μας φέρνει ακόμη πιο κοντά από πλευρά της Λετωνικής Προεδρίας. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Βίξτρομ και τους συναδέλφους της διότι ήταν καλοί ε, διαπραγματευτές μαζί μας. Ευχαριστώ την Επιτροπή και ιδιαίτερα τον κύριο Άιντενμπεργκ για όλη την εργασία και εμπειρογνωμοσύνη για το τεχνικά περίπλοκο αυτό θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. And, uh, we go... Οπότε να περάσουμε τώρα στην έκθεση της κυρίας ε, Ρέντα. Λοιπόν, να ξεχνήσουμε την τροπολογία 113 υπέρ. 130 συγγνώμη. Υπέρ. Επαναλαμβάνω. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ. Αποχές λέει ο πρόεδρος. Α, με κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 1. 1 για την παράγραφο 1D υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Εγκρίνεται. 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 150 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. παράγραφο 2α ήτρε 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Still missing somebody. Παρακαλώ, ε, κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ήμικο 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 165. Για την παράγραφο 2b. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Doesn't work. Yes, we are checking. Ναι, να κάνουμε έλεγχο. Τις 166. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τα μηχανήματα ψηφοφορίας. Υπάρχει τεχνικός. Do we have a technician here? Τεχνικός εδώ παρακαλώ. Well, let's try to do it manually. Um, Ωραία, θα επιχειρήσουμε διανατάσσεως της χειρός. 166. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Μπορεί κάποιος να μετρήσει. Εννέα κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Εκατόν εξτρεφτό. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 169. Υπέρ. κατά, αποχές, εγκρίνεται. 170 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 172 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 175 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 176. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 177. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 189. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 190. Υπέρ. Κατά. Σηκώστε το χέρι παρακαλώ, Είστε κατά. Μάλλον από την αρχή. Ας αρχίσουμε από την αρχή. Υπέρ. Κατά. Δέκα. Συγγνώμη. Ας προσπαθήσουμε τώρα ηλεκτρονικά. Λειτουργεί.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 διότι τα μηχανήματά σας, τα δικά σας, δουλεύουν. Είμαστε στην τροπολογία 190. του κυρίου Φως. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Ποιοι είναι κατά. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. 12 υπέρ, 11 κατά. Αποχές. Εκατόν ενενήντα οχτώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκατόν ενενήντα εννέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 200. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 201. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ποιος είναι υπέρ από το Προεδρείο. Δύο. Και κατά. Τρεις. Απορρίπτεται λοιπόν. τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος και εδώ. Και σε εμείς το Προεδρείο. Ποιοι είναι υπέρ, τρεις Ποιοι είναι κατά, δύο. Απορρίπτεται. Λοιπόν, είμαστε στην τροπολογία 203. Εγκρίνεται. 204. voting, yeah. 25 people, no, 25 cards. 26 cards in, but 25 people voted. Mrs. Reda. Κύριε Ρέντα, θα μπορούσαμε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία και να διασφαλίσουμε ότι ψηφίζει ο σωστός αριθμός, γιατί νομίζω υπάρχει ένας υπεράριθμος.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 the person that does not vote. Κάποιος δεν ψηφίζει και ωστόσο χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική του κάρτα. Μάλιστα, ωραία. Εγκρίθηκε λοιπόν. 204, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ηλεκτρονικός έλεγχος. Απορρίπτεται. 206. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 207. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 225. Υπέρ. 225. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Απορρίπτεται. τριάντα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 232. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 233. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.34 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Απορρίπτεται. 2.35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 266 σχετικά με την παράγραφο 6α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 280. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 283 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 284 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 18 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 288. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 9. Υπάρχει κάποια προφορική τροπολογία. Παρακαλώ. Η προφορική τροπολογία λοιπόν θα προσθέσει after swift ratification και χωρίς να γίνεται η έγκριση υπό προϋποθέσεις ε, Αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Νομικού Πλαισίου. Εγκρίθηκε λοιπόν 306 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 222 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Εγκρίνεται. Μάλιστα, αλλιώς μας φαινόταν εδώ στο Προεδρείο. 323. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 324. Υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. 325 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 326 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 245. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 246. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 348. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 350. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Εγκρίνεται. 3.51 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 351 λοιπόν, πρώτο τμήμα. Μας λείπουν 3. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 352. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 353. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 355. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για την 355. Απορρίπτεται. 356. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 363. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος. Απορρίπτεται. Τρία Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 365. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 366. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. «389 ηλεκτρονικά». Απορρίπτεται. 396 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 411 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 412 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 414 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος απορρίπτεται 418 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 419 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 421 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 429. Υπέρ. Με συγχωρείτε. 4.29 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Αγκρίνεται. 430. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 451 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 471. Υπέρ. Κατά. Και ηλεκτρονικός έλεγχος. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 476. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 476. Εγκρίνεται. 487. Υπέρ. Κατά. 487. Καταπίπτει. Ήτρα 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 507 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 508 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 509 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 523 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 524 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 525 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 525. Απορρίπτεται. 526. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 527. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 528. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Απορρίπτεται. Ήμκο 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 23 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχο για το πρώτο τμήμα. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 532 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 538 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 539 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5.53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας την ελέγξουμε. Ξέρω ότι είναι κουραστικό, αλλά σας παρακαλώ να σηκώνετε καθαρά τα χέρια σας. Εγκρίνεται. 5.54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγγνώμη. Εγκρίνεται. 5.55 υπέρ. Α, με συγχωρείτε. 554. Τι. Ο, ο, 5 556, δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε το πρώτο τμήμα. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήτρα 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΥΜΚΟ 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται Επτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 26 υπέρ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 εγκρίνεται 43 υπέρ κατά <clears throat> αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε ωραία ελέγχουμε τις 44 Άλλος ένας παρακαλώ. Εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ανέλεξουμε. Ωραία. Ελέγχουμε την 69. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Θα την έλεγξουμε. Ελέγχουμε την 71. Εγκρίθηκε. 75 υπέρ. Συγγνώμη, συγγνώμη. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε το 74. απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 76 υπέρ κατά αποχές έλεγχος της 76 εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται να την ελέγξουμε την 94 απορρίπτεται 101 υπέρ. Α, α καταπίπτει. 104. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Έλεγχος της 104. Απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε 107. Απορρίπτεται. Συμβαστική 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το σύνολο του ψηφίσματος. Εγκρίθηκε.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 Πρέπει να επιστρέψουμε στις ε, μία ψηφοφορία για κάθε έκθεση. Μήπως μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτών, γιατί ψηφίζουμε τόση ώρα αν έχουμε χρόνο κύριε Πρόεδρε. Υποστηρίζει κανείς ε, αυτό το αίτημα. Δεν νομίζω. Οπότε συνεχίζουμε. Περνάμε στην αναφορά υπαρισμών 0486 κάθετος 2014 ηλεκτρονικός I close the Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Μία ακόμη που είναι η νομική βάση προστασία από τις συνέπειες εξοεδαφικής εφαρμογής νόμων που θεσπίστηκαν από τρίτη χώρα. Μία ακόμη φορά ηλεκτρονικός. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Πάμε στο σημείο 20, μια ακόμη νομική βάση, για την πρόταση οδηγίας για τους ναυτικούς, που τροποποιεί τις οδηγίες 2008-94 μεταξύ άλλων έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τώρα ε, περνάμε στις κωδικοποιήσεις. Η συγγητής είναι ο κύριος Μαστάλκα, έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. ακόμη κωδικοποίηση πάλι του κυρίου Μαστάλκα. Ένα ψηφοφορία είναι κατά τη σημειογόνου τιμολόγηση των πλοίων. Εγκρίνεται. Και αυτή. Ωραία. Η κυρία Κάουφμαν μήπως θέλει να πάρει το λόγο πριν περάσουμε στην ψηφοφορία τη εκθεσή τη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις για τον κατάλογο ψηφοφοριών γιατί ορισμένες συνάδελφοι μπορεί να μην έχουν το σωστό κατάλογο. Το πρώτο αφορά τη συμβαστική 5. Αν εγκριθεί στην αρχή η πρώτη ψηφοφορία τότε πρέπει να ψηφιστεί η 39 και όχι η 37. Και δεύτερον, έχουμε δύο ταυτόσιμες τροπολογίες, ΙΜΚΟ 23 και NV90 και αφορούν την, την παράγραφο 18 σε 28 και όχι για το 11α. Αλλά νομίζω ότι έχετε ήδη λάβει αυτή την πληροφόρηση. Ich soll Θα τα ξαναπώ. Λοιπόν, τα ξαναλέω. Με συγχωρείτε συνάδελφοι, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να τα διατυπώσουμε όλα ακριβώς. Λοιπόν, πρώτον, η πρώτη ψηφοφορία, συμβαστική 5, εάν εγκριθεί, τότε θα πρέπει να ψηφίσουμε την 39, όχι την 37. Και δεύτερον, Έχουμε δύο ταυτόσημες. ΙΜΚΟ 23 και ΕΜΒΙ 39 αφορούν την παράγραφο 18C και άρα στη σελίδα 20 όπως έχω εδώ μπροστά μου το κατάλογο και όχι την παράγραφο 11α. so please control us that we proceed. Μάλιστα, ωραία. Οπότε θα συνεχίσουμε υπό τον έλεγχό σας. Να αρχίσουμε με τη συμβαστική τροπολογία 5, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ, τη 41. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος νομίζω ότι απορρίπτεται απορρίπτεται όντως Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Γκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές παρακαλώ να το ελέγξουμε και αυτό ηλεκτρονικώς εγκρίνεται τροπολογία 60 υπέρ κατά Ας την ελέγξουμε κι αυτή γιατί δεν είμαι βέβαιο. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήμκο 5, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. NV16, ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται MV30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται MV40 υπέρ κατά αποχές έλεγχος Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά καλύτερα να ελέγξουμε Απορρίπτεται. όντω. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 74. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 75. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Έλεγχος της 79. Απορρίπτεται. 78. Υπέρ. Κατά. Να την ελέγξουμε, αλλά νομίζω ότι απορρίπτεται. Απορρίπτεται όντως. Συμβιβαστική τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την ελέγξουμε, παρακαλώ. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 87 υπέρ κατά να, να ελέγξουμε καλύτερα την 87 Εγκρίνεται. Δεν μου φαινόταν τόσο βέβαιο. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχέρ, εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχέρ, απορρίπτεται. 93. Ναι, όχι 93 όχι την 93, 95 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο... Α, όχι, δεν την ψηφίζουμε αυτή, λέει ο πρόεδρος. Ψηφίζουμε την MV23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκατόν εννέα. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο παρακαλώ απορρίπτεται συμβιβαστική 19 τρία τμήματα Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Παρακαλώ έλεγχος. Ξέρω, είστε κουρασμένοι. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ένδυ 12. Παράγραφος 13α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 20. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 120, συγγνώμη, τροπολογία 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 129 όχι, 128, 128 διευθύνει ο πρόεδρος, υπέρ, Νέα διόρθωση 129 τελικά. Γιατί καλύπτεται η 128 από, τον, ε, από τη συμβιβαστική. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για να μην υπάρχουν ε, αμφιβολίες, ας ψηφίσουμε και την 128. Εντάξει, λοιπόν, υπέρ της 128. Κατά. Έλεγχος. Απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Εγκρίνεται. Κύριε Γάφμαν. Ναι, να σας πω ότι η τροπολογία 129 είχε συνταχθεί στα αγγλικά και η γερμανική μετάφραση έχει πάρα πολλά λάθη. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις άλλες γλώσσες, αλλά με τα γερμανικά έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να το κοιτάξουμε, να ψηφίσουμε αν γίνεται μόνο το αγγλικό πρωτότυπο της τροπολογίας. So we one yes. One Okay. Uh, we vote on one Να ψηφίσουμε την 130. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά έλεγχος. Εγκρίνεται. 143. Υπέρ. So it falls. One for one. Λοιπόν, 141 καταπίπτει. 141 is incompatible with Η 141 δεν είναι με την 139. Οπότε θα ψηφίσουμε την 143. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 144. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 145. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Εγκρίνεται. 146. Υπάρχει προφορική τροπολογία. Όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 147. Υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 150 υπέρ κατά έλεγχος Εγκρίνεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά. Ξανά. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 163. Α, όχι, όχι. Employment 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 168 υπέρ κατά αποχές έλεγχος Απορρίπτεται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ. Έλεγχος. Απορρίπτεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Employment 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος έλεγχος της 192 εγκρίνεται 194 με συγχωρείτε. 195 υπέρ. Εκατόν Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κύριε Κάουφμαν, πρέπει να πάμε στην τροπολογία 206. Να ψηφίσουμε τη 206 και μετά να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ. 206. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Απορρίπτεται. 208. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 209. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 210. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 224. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 225. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1.19. 19. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Εγκρίνεται. 2.28 υπέρ κατά Α, καλύπτεται. Ωραία, προχωράμε. Employment 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Employment 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Employment 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Employment 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Employment 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Employment 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Employment 35 υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. Ίμκο 4 υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. Ινκο 21 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. ίνκο 21. Απορρίπτεται. Ίμκο 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήμκο 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ένβι 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ένβι 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ένβι 25. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. NV26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. NV27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. NV28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. NV32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. NV33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33, NV33, ηλεκτρονικός έλεγχος. Εγκρίνεται. μαλιστα με Εκπλήσωμε. NV34. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. NV37, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5, υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τροπολογία 5. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε λοιπόν τελική ψηφοφορία. Η ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται συγχαρητήρια κυρία Κάουφμαν.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 and the floor goes to the rapporteur, uh, Mr. De Grandes Pascual. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της ε, Επιτροπής και του Συμβουλίου, και όλοι όσοι παρακολουθούν αυτό το τόσο συναρπαστικό θέμα που πρέπει να παρακολουθήσουν τη συζήτηση για το τόσο επίμαχο θέμα. Επανέρχεται στην Επιτροπή μας η πρόταση οδηγίας για τις μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με τα αρχικά SUP, SUP. Θεωρητικά αγαπητοί συνάδελφοι, εάν όλα ήταν καλά ή τουλάχιστον φυσιολογικά, θα συζητούσα μια έκθεση του εισηγητή. Αλλά δεν έχουμε σήμερα τις συνθήκες για να θεωρήσουμε ότι ε, λειτουργούμε σε ομαλές συνθήκες. Είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις. Και Όταν ε, όμως εγώ ε, αποφάσισα να αναλάβω αυτό το θέμα δεν έλεγξα αν στην πισίνα είχε νερό ή αν θα σπάγαμε τα μούτρα μας πέφτοντας. Αλλά ας έχουμε, όπως είχα και εγώ, θετική στάση. Αλλά με την αναγκαία ε, προφύλαξη. Έχουμε μια πρόταση της Επιτροπής που μπορούμε να τη βελτιώσουμε, να καταλήξουμε σε μια διατύπωση που να έχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Με βάση αυτές τις προποθέσεις άρχισα να εργάζομαι και έλεγξα την πολιτική θερμοκρασία των επιτρόπων, των, του κλάδου και γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα να αναβάλω την υποβολή έκθεσης και να υποβάλω ένα σχέδιο εργασίας για να δούμε ποια είναι τα προβλήματα και ποιες οι δυνατότητες υπέβαλα αυτό το κείμενο, υπήρξε ανοιχτός διάλογος με τους συναδέλφους στην Επιτροπή και χρειάστηκε να αναβάλω εκ νέου την υποβολή της έκθεσης. Ομολογώ ότι όλο το χρόνο που είχα για να μιλήσω με την Επιτροπή, το Συμβούλιο, με τις πολιτικές ομάδες, με όλους τους ενδιαφερομένους, κατάλαβα ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε με το στόχο της έκθεσης. Να βελτιώσουμε δηλαδή τη δυνατότητα των μικρομεσαίων να ε, τη δυνατότητα των μικρομεσαίων να έχουν πρόσβαση στην αγορά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι συμμεριζόμεθα τον τρόπο. Σήμερα έχουμε ένα νέο στοιχείο όμως ενώπιόν μας. Είναι η θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 28 Μαΐου, που έχει μεγάλη σημασία. Όποιος παρακολουθεί προσεκτικά αυτά τα θέματα, διαπιστώνει ότι υπάρχουν διχόνες και εντός του Συμβουλίου Φυσιολογικό θα πει κανείς. Αλλά υπήρχαν διάφορες δυσχέρειες. Κάποια στιγμή υπήρχε μια μειοψηφία που είχε μπλοκάρει το θέμα κατόπιν ε, ξεπεράστηκε αυτό. Σήμερα έχουμε την επίσημη θέση. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι το Συμβούλιο έρχεται με πολλή αποφασιστικότητα αλλά θα πρέπει να προσέξουμε τι θα πούμε για το πώς αναλύουμε τη θέση του. Οπωσδήποτε το Συμβούλιο με τη θέση του τροποποιεί πολύ την άποψη της Επιτροπής. Κατά 60% το κείμενο του Συμβουλίου διαφέρει από το κείμενο της Επιτροπής, αλλά δεν επιλύει μερικά θέματα που είχαν τεθεί από την αρχή. Για παράδειγμα, πώς θα καταπολεμήσουμε το dumping, το κοινωνικό dumping, πώς θα καταπολεμήσουμε το ενδεχόμενο ο καθένας να διαλέγει τη δικαιοδοσία που προτιμάει. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να επιληθούν. Αν θέλουμε πραγματικά να συνδυάσουμε τις θέσεις των μεν και των δε για να προχωρήσουμε. Επιπλέον. τίθεται ένα αμφιβόλο εάν και κατά πόσο υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε αυτή την πρόταση. Αυτό είναι βασικό θέμα. Δεν θέλουμε να κάνουμε θεωρητικές προσπάθειες. Είμαστε νομοθέτες και γι' αυτό έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Επίσης, το Κοινοβούλιο έχει επίσης δώσει γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης που απέρριψε την πρόταση τη Κομισιόν. Και επίσης η Επιτροπή Εσωτερικού Εμπορίου δεν καταφέρνει να καταλήξει σε πλειοψηφίε για να εγκρίνει τις θέσεις της. Θέσεις που να συμφωνεί με αυτές και ο εισηγητή. Άρα υπάρχει ενδεχόμενο ο εισηγητή τελικά να απορρίψει τη γνωμοδότηση αυτή. Σας περιγράφω λοιπόν την κατάσταση όπως είναι. Γιατί στην πολιτική δεν πρέπει να γελιόμαστε, πρέπει να είμαστε σοβαροί, να επιχειρούμε να καταλήξουμε σε λύσεις, να υπερβούμε τις δυσχέρειες. Έχουμε πολλές δυσχέρειες και εδώ ως νομική επιτροπή, γιατί στις προηγούμενες συζητήσεις νομίζω ότι κατέθεσαν σαφείς. Ελπίζω λοιπόν ότι θα καταστούν επίσης ε, σαφείς. Αλλά υπάρχει ένα νέο στοιχείο, όπως είπα η θέση του Συμβουλίου. Οπότε θα άξιζε τον κόπο να μπούμε στην ουσία. Οπότε, η κατάσταση είναι δύσκολη, είναι λοιπόν αναγκαίο να ακούσουμε σήμερα, σήμερα το Συμβούλιο για να δούμε ποιες είναι οι γενικές του κατευθύνσεις για τη ΣΟΥΠ, να ακούσουμε την Κομισιόν, να δούμε πώς ε, αντιμετωπίζει αυτές τις αλλαγές στην αρχική της πρόταση και να ακούσουμε και την ε, δική μας απόψη εδώ των συναδέλφων. Αυτό νομίζω εισαγωγικά έπρεπε να πω. Θα προτιμούσα να κάνω μια εισαγωγή, να σας πω αλλά πριν κάνω την εισαγωγή, καλύτερα να ακούσω την Επιτροπή και το Συμβούλιο, να ακούσω τους συναδέλφους και εγώ ως περιμένω βέβαια να λάβω το λόγο στο τέλος για να αποτιμήσω πώς έχουμε προχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γουίνα Μπάιτερε από το ε, Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, πολύ καλά το είπατε το όνομά μου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε ε, Σφομπόντα που μου δίνετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Ε, Γκούνα Πάιντερε είναι το όνομά μου και είμαι η επικεφαλής ε, ε, του Λετωνικού ε, Μητρώου Επιχειρήσεων και επίσης είμαι και πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Συμβούλου που ασχολείται με το θέμα των εταιριών αυτών. Θα ήθελα εκ μέρους της Λετωνικής Προεδρίας να σας ενημερώσω σε σχέση με την γενική προσέγγιση μας για το θέμα αυτό. Ε, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στις 28 Μαΐου. Ε, δεν είναι εύκολο ποτέ να υπάρχει συμβιβασμός. 14 ε, συνεδριάσεις χρειάστηκαν ε, υπό την ελληνική, ιταλική και Λετωνική προεδρία για να ολοκληρωθεί το κείμενο και κατά τη διάρκεια των ομάδων εργασίας υπήρξαν πολλές ανησυχίες που εκφράστηκαν από τις αντιπροσωπείες μεταξύ των οποίων υπήρχαν και κάποιες που έμοιαζαν σε μεγάλο βαθμό με αυτές που εκφράσατε κι εσείς εδώ στη συνεδρίαση της Επιτροπής σας. Καταφέραμε βέβαια να καταλήξουμε σε συμβιβασμό ε, εστιαζόμενοι σε δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι η ε, ηλεκτρονική ε, εγγραφή καταχώρηση των εταιριών, ε, των εταιριών αυτών που κατά τη γνώμη μας θα είναι επωφελές για, το, για την ψηφιοποίηση στο μέλλον και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο Υπουργό Οικονομικών μας που είπε κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητάς μας ότι έχουμε εδώ μια μεγάλη ευκαιρία και από πρακτής και από συμβολικής απόψεως να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να ψηφιοποιηθούν περισσότερο για να, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καταχωρούνται ηλεκτρονικώς. Υπάρχει βέβαια και η πρόκληση, υπάρχουν διάφορες προκλήσεις ε, που αφορούν κυρίως τη διασυνοριακή αναγνώριση. Επομένως, ε, ε, υποχρεούνται βάσει του συμβιβασμού τα κράτη-μέλη να ε, κάνουν τέτοιου είδους αναγνώριση όταν υπάρχει ε, συμβιβασμός με τον, ε, με τον κανονισμό που διέπει τις εταιρείε αυτές. Επίσης, όσον αφορά τη διευκόλυνση της σύσταση εταιρείων, κυρίως για τις νεοσύστατες εταιρείε και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις θηγατρικές τους, πιστεύουμε ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη. Ε, θεωρούμε ότι πρέπει να μειώσουμε την δυνατότητα καταχρήσεων, ε, δηλαδή να ε, προσπαθήσαμε να, να, να, να, υπάρχει, να υποχρεώσουμε τις εταιρείες να έχουν έναν ισορροπημένο ισολογισμό πριν από τη σύστασή τους και πιστεύουμε ότι ο κίνδυνος για αυτές τις εταιρείες δεν είναι υψηλότερο σε σχέση με άλλες μορφές εταιρείων που υπάρχουν ήδη. Επομένως, συμβιβαστικό κείμενο συνιστά ε, προστιθέμενη αξία σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση γιατί επιτρέπει μια απλή σύσταση εταιριών, κάτι το οποίο θα είναι πολύτιμο σε ε, διασυνοριακές περιπτώσεις. Ε, θα ζητούνται βέβαια ελάχιστε πληροφορίε από του ιδρυτέ, και οι περισσότερε πληροφορίε θα παρέχονται από το κράτο. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντα ότι μα ε, χαροποιεί όλο ιδιαίτερο ο συμβιβασμό που καταφέραμε, στον οποίο καταφέραμε να καταλήξουμε στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα, γιατί η ψηφιακή Ευρώπη και η ανταγωνιστική Ευρώπη είναι δύο από τι προτεραιότητε μα. Όμω, ε, η Προεδρία μα πλησιάζει προ το τέλο τη. Ε, και είναι εδώ η κυρία Ελένη Μασάρ, η οποία θα είναι η πρόεδρος του φακέλου αυτού, επικεφαλής του ε, φακέλου αυτού ε, κατά την ε, Προεδρία του Λουξεμβούργου, οπότε θα σας ενημερώσει και εκείνη εντάχει για τις προτεραιότητες της Προεδρίας του Λουξεμβούργου για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Χέλεν Μασάτ από στο Υπουργείο Οικονομικών του Λουξεμβούργου. Είμαι μέρος της ε, διαπραγματευτικής ομάδας και να σας πω ότι ως ε, επερχόμενη Προεδρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Λετωνική Προεδρία για την εξαιρετική δουλειά και πρόοδο που έχει κάνει σε αυτό το θέμα. Παρά την ε, μεγάλη συνένεση των κρατών μελών για τους ε, γενικότερου στόχους της πρόταση αυτής, τη διευκόλυνση δηλαδή και ενθάρρυνση, δημιουργία δημιουργίας μονοπρόσωπων εταιριών περιορισμένης ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Λετωνική Προεδρία ωστόσο έπρεπε να καταβάλει ιδιαίτερε προσπάθειες και δεσμεύσεις έτσι ώστε να επιλύσει τα εκκρεμή ζητήματα. Η επερχόμενη Προεδρία θεωρεί πως η γενικότερη προσέγγιση της Ελαττονικής Προεδρίας είναι μια πάρα πολύ καλή βάση και ελπίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, ψηφίσει ε, σχετικά όπως ε, προέβλεπε. Αναμένουμε με χαρά της, την καλή συνεργασία με το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να επιτευχθεί μια σωστή και πλήρη συμφωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Χόγερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω ενώπιον της Επιτροπής αυτής. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και οι απόψεις που έχουν ακουστεί είναι πολλές. Τους τελευταίους μήνες έχουμε ακούσει πάρα πολλά ότι πρόκειται για ξέπλυμα χρήματος, για κοινωνικό τάμπινγκ, για εταιρείε που είναι πλασματικές, για φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή. Και πραγματικά πρέπει να αναρωτηθούμε πώς είναι δυνατόν το Συμβούλιο να έχει ψηφίσει για κάτι τέτοιο, για όλα αυτά, με ειδική πλειοψηφία. Θα σας δώσω ορισμένα στατιστικά στοιχεία που στηρίζουν την πρόταση αυτή. Καταρχάς, δεν υπάρχει καμία πρόταση που να είναι απαλλαγμένη από τον οποιονδήποτε κίνδυνο. Πρέπει να εντοπίσουμε την προστιθέμενη αξία και τις ασφαλιστικές δικλείδες που μπορούμε να έχουμε στην διάθεσή μας. Επιπλέον, δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Ελευθερία εγκατάσταση, διασυνοριακέ δραστηριότητε προ το συμφέρον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, αυξήσει την, ε, το δυναμικό τη και να αυξήσει την δυνατότητα ψηφιοποίησης, ε, να δοθεί η δυνατότητα διασυνοριακής διαδικτυακή. Καταχώρηση των εταιριών που θα ενισχύσει την ενιαία αγορά. Επίσης, η πρόταση αυτή θα συνεισφέρει στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης, διότι όπως ξέρετε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 95% των εταιριών περιορισμένης ευθύνη στην Ένωση. Επίσης, με τους ε, μετόχους Επίση, ε, το SGP δεν θα έχει μειοψηφούντε σε θα έχει μόνο έναν μέτοχο. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά πλεονεκτήματα, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ευκαιρία που μας έδωσε να δημιουργήσουμε δημιουργικές λύσεις για ε, το εταιρικό δίκαιο. Η ανάγκη για ένα τέτοιο μέσο έχει επιβεβαιωθεί από πολλούς φορείς, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από μη κυβερνητικέ οργανώσεις και από νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι τόσο καλά οργανωμένες όπως ε, οι μεγαλύτερες εταιρείες. Έχουν λίγα μέσα στη διάθεσή τους και η φωνή τους δεν γίνεται ιδιαίτερα ακουστή στις Βρυξέλλες. Είναι όμως εξίσου σημαντικές. Υπάρχει μεγάλη προστιθέμενη αξία στην πρόταση, διότι αφορά την εναρμόνιση βασικών κανόνων που θα διέπουν τη λειτουργία των μονοπρόσωπων εταιριών. Θα διευκολύνει λοιπόν τις ε, επιχειρήσεις αυτές, ιδιαίτερα στην περίπτωση που θέλουν να δραστηριοποιηθούν διασυνοριακά. Ας δούμε τώρα τους κινδύνους. Όπως είπα, υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν κίνδυνοι. Πρέπει να τους εντοπίσουμε, να τους πάρουμε στα σοβαρά και να βρούμε λύσεις. Όμως, ας κάνω μια σύγκριση με ένα αυτοκίνητο. Όταν σχεδιάζουμε ένα νέο αυτοκίνητο, φυσικά και λαμβάνουμε υπόψη τους κινδύνους και τα πιθανά ατυχήματα. Η λύση όμως δεν είναι να σταματήσουμε το σχεδιασμό του νέου αυτού τύπου αυτοκινήτου. Η πρόκληση είναι και να σχεδιάσουμε το αυτοκίνητο και να το κάνουμε όσο το δυνατόν ασφαλέστερο. Τώρα για το ηλεκτρονικό μέσο θα υπάρχει μία διαδικτυακή αίτηση. Όπως για παράδειγμα όταν κάνω αίτηση για το γιο μου στο πανεπιστήμιο. Θα μας ε, γλιτώσει χρόνο και χρήμα. Όλες αυτές οι αιτήσει θα γίνονται χωρίς την ανάγκη συμβολιογράφου ηλεκτρονικά. Και τώρα κάτι που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό. Έχουμε συμπεράνει ότι η ηλεκτρονική εγγραφή, καταχώρηση, είναι ένα σύστημα πιο δύσκολο, πιο εκλεπτισμένο και πολύ πιο δύσκολο να ε, γίνει αντικείμενο κατάχρησης. Τώρα, άλλες ανησυχίες, εάν θα επιδεινωθούν τα κοινωνικά πρότυπα και αν θα ευνοηθεί το κοινωνικό dumping. Φυσικά και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το αποφύγουμε. Όμως, να σας πω ότι οι κοινωνικές πτυχές ρυθμίζονται από άλλη ευρωπαϊκή νομοθεσία και η πρόταση για τις SUP γίνεται με κάθε επιφύλαξη προς αυτές. Προς τον κοινωνικό τομέα. Επίσης, γίνεται μια αναθεώρηση αυτήν την ε, περίοδο για την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων και το ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο πρέπει να συνάδει με την ανάπτυξη και την εξέλιξη στην αγορά έτσι ώστε να αποφευθεί το κοινωνικό dumping. Αυτό το δηλώνει η Επιτροπή ξεκάθαρα. Επίσης, εάν θα οδηγήσει σε περισσότερη φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή η πρόταση αυτή, να σας πω ότι το Συμβούλιο έχει διαγράψει τελείως το, την αναφορά στην έδρα. Δηλαδή θα διατηρηθεί το status quo, δεν θα αλλάξει τίποτα. Τα κράτη-μέλη θα έχουν την πλήρη ελευθερία να ε, ρυθμίσουν την, ε, τις έδρες μιας επιχείρησης. Την έδρα ή τις έδρες. Και τέλος, καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Υπάρχει ένα εφιστάμενο πλαίσιο, εγκεκριμένο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τρεις εβδομάδες. Η πρότασή μας είναι 100%, 120% σύμβατη με την οδηγία για την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Διότι ο κύριος δικαιούχος πρέπει να ταυτοποιείται κατά τη διάρκεια της ε, εγγραφής. Τέλος, να τονίσω κύριε Πρόεδρε ότι παραμένει ένα μέσο του εταιρικού δικαίου. Το Συμβούλιο σίγουρα μπορεί να κάνει περισσότερα και αυτή η Επιτροπή, η δική σας Επιτροπή μπορεί να κάνει περισσότερα. Έργο σας είναι να αντιμετωπίσετε τις ε, κρεμίσει ανησυχίες και να μειωθεί η γραφειοκρατία στην ε, καταχώρηση μονοπρόσωπων εταιρείων για το συμφέρον όλων μας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Νίμπλερ, ζητήσατε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να συγχαρώ τον εισηγητή μας, όχι μόνο για αυτή την έκθεση. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό πώς ε, φρόντισε να συμμετάσχουμε όλοι με ένα έγγραφο εργασία που μας παρουσίασε τα θέματα με λεπτομέρεια και τώρα έχουμε τα τελευταία στοιχεία με τη θέση κατά πλειοψηφία του Συμβουλίου νομίζω ότι είναι θαυμάσια συνεργασία και ευχαριστώ ιδιαίτερα ως Επιτροπή επανειλημμένα είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε το θέμα και καταρχάς δεν θέλω ε, να σας κρύψω ότι είμαι ιδιαίτερα επικριτική. Ο συγητής μας σωστά είπε ότι βεβαίως ε, καταρχάς θετική αλλά ε, και ιδιαίτερα επιφυλακτική διότι στόχος μας ήταν να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες να μπορούν να έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα. Συμμερίζουμε αυτή την άποψη και εν ώψη της ε, ψηφιοποίησης, αλλά παρόλα αυτά έχω πολλές αμφιβολίες για το εάν και κατά πόσο αυτή η πρόταση θα επιτύχει αυτούς τους στόχους. Και όταν ακούω τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, ο οποίος είναι σαν να μας λέει ότι ε, άμα δεν δεν κερδίζεις και τίποτα. Νομίζω ότι από τις εμπειρίες που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια και τις δεκαετίες τελικά δεν έχουμε μάθει τίποτα και για να τα πω και πολύ προσεκτικά είχαμε, έχουμε όπως ξέρετε δημιουργήσει μια ειδική επιτροπή για φορολογικά θέματα στο Κοινοβούλιο. Πώς είναι δυνατόν να μας λέτε ότι πολύ γρήγορα, χωρίς γραφή και να μας λέγεται ότι οι κίνδυνοι δεν είναι τόσο σημαντικοί. Ε, δεν ξέρω εάν αυτά δεν ανησυχούν την Κομισιόν αλλά εμείς όταν θα πρέπει να πάμε στους ψηφοφόρους και να πούμε τι επιτρέπουμε για να διευκολύνουμε το τη διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα, τότε θα ε, δραστηριότητα θα μας πούνε μα πώς διαπιστώνετε πού φορολογείτε και τι φορολογείτε και βεβαίως και κάποιος άλλος συναλλασσόμενος θα πρέπει να ξέρει με ποιες εταιρείε συναλλάσσεται και αν δεν μπορεί να είναι, υπάρχει κάποιο ένα μητρό ε, ξέρετε ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη σε ένα τέτοιο μήτρο. Δεν είναι το να μα λέτε ότι υπάρχουν κίνδυνοι αλλά πρέπει να του αντιμετωπίζουμε, να του αναλαμβάνουμε. Δεν μπορώ να αποδεχθώ τέτοιε διατυπώσει. Αναφέρθηκα επίση στο γεγονό ότι μπορεί να επιδιώκουν να βρουν την καλύτερη δικαιοδοσία, το forum shopping. Και επίση για το αρχικό κεφάλαιο αυτών των ZUP. Πώ θα διαπιστώσουμε, πώ θα εσφαλίσουμε ότι θα είναι στη διάθεση τη εταιρεία και ότι αυτή η εταιρεία όταν έρχεται σε επαφή με τρίτους και συναλλάσσεται είναι αξιόπιστος εταίρος. Αυτές οι προτάσεις ούτως ή άλλως στην αρχική πρόταση της Κομισιόν δεν ήταν αρκετές για μένα και για το Forum Shopping βλέπω ότι διαγράφησαν όλες οι διατάξεις γι' αυτό και δεν μπορώ να το υποστηρίξω αυτό για το πώς θα διαπιστώνουμε ποια είναι η εταιρεία, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ποιος είναι ο ιδρυτής. Δεν έχει επιληθεί ακόμη να δούμε αν θα γίνει τίποτα γι' αυτό, να δούμε τι θα υπάρξει, αλλά γενικά να πω, νομίζω ότι ε, έχει μεγάλη σημασία η αξιοπιστία των δημοσίων μητρώων επιχειρήσεων. Βεβαίως θέλω να αξιοποιήσουμε την εσωτερική αγορά, αλλά πρέπει να υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας. Αν δεν υπάρχουν για αυτή τη νέα μορφή εταιριών, πρέπει να το ξανασκεφτούμε επιχειρούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δημιουργήσουμε κάτι το καινούριο με νέους κανόνες αλλά αυτά τα σουπ δεν είναι το είδαμε και με το Σοσιατάς Ευρωπαία δεν ισχύει πρόκειται για εθνικές μορφές <clears throat> και τα 28 κράτη-μέλη μπορεί να ερμηνεύσουν διαφορετικά το νομοθέτημα αυτό και θα θεωρούνται όλα αυτά σουπ αλλά δεν θα είναι τα ίδια Άρα λοιπόν όσοι θεωρούν ότι είναι προστιθέμενη αξία αυτή η πρόταση πρέπει να το ξανασκεφτούν. Δεν μπορούμε να πούμε, κοιτάξτε να δείτε, ναι υπάρχει κίνδυνος αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω οι διερμηνείς να έχουν λίγη ακόμη υπομονή. Ο κύριος Φως. Βος. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ε, εισηγήτρια για αυτήν την πάρα πολύ προσεκτική προσέγγιση. των εισηγήτη με ε, Τώρα, η Αγγέλικα Νίμπλελ έχει ήδη εκφράσει κάποιες ανησυχίες που συμφωνώ και εγώ και το Συμβούλιο να πω ότι έχει κάνει μεγάλες αλλαγές στην πρόταση. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Προεδρία του Συμβουλίου εάν υπάρχει σήμερα, αυτή τη στιγμή, μια πλειοψηφία για αυτή ε, την ε, πρόταση, διότι ακούγονται φήμες ότι κάποιες ε, χώρες έχουν δισταγμούς. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω αν σήμερα, σήμερα που μιλάμε, υπάρχει συμφωνία. Εμείς έχουμε αντιληφθεί αυτήν την μεγάλη ασάφεια που υπάρχει και αυτήν την ανασφάλεια. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να προτείνω να εισαγάγουμε ένα μια διαφορετική διαδικασία όπου να είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε και να ανακοινώνουμε το ε, στο κοινό αποφάσεις όταν αυτές θα έχουν ληφθεί και, και όχι όσο ακόμα υπάρχει αβεβαιότητα. Έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος να γίνονται όλες οι τροποποιήσεις ή οι αλλαγές για να μπορούμε και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δούμε τι γίνεται. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν άτυπο τριμερή διάλογο, για παράδειγμα, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με το εκάστοτε θέμα, με το συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να συμφωνούμε, να διαφωνούμε με κάτι. Προτού όμως γίνονται ανακοινώσεις προς τα έξω. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους εμπλεκόμενους να αναλογιστούν αυτή την πρόταση και να προτείνω και στον εισηγητή να βρει μια πρόταση η οποία θα δίνει λύση για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Επίσης, έχετε απόλυτο δίκιο όταν λέτε πως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή και σας ευχαριστώ πολύ που το αναφέρατε και εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Τέσσερα λεπτά ακόμη έχουμε στη διάθεσή μας με τους διερμηνείς. Οπότε θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Ντεγκράντες να μας πει ορισμένα πράγματα πώς πιστεύει ότι πρέπει να εγγράψουμε το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη επόμενη συνεδρίασής μας και μήπως η κυρία Ρέγνερ μεταξύ μπορεί και εκείνη να μας πει κάτι γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα κάνω μια πάρα πάρα πολύ σύντομη δήλωση να πω ότι φαίνεται ότι ούτε στο Συμβούλιο είναι σαφή τα πράγματα. Δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη απόρριψη ή έγκριση της πρότασης αυτής. Και παρατήρησα ότι όντως υπάρχουν μεγάλες αμφιβολίες και στο Συμβούλιο και πιστεύω πως ε, οι αμφιβολίες αυτές δεν έχουν ακόμα επιληθεί. Αμφιβολίες σχετικά με τη χρηματοδότηση, με την τρομοκρατία, με την συμμετοχή των εργαζομένων, με την φοροαποφυγή, με το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης. Παραμένουν λοιπόν αυτά τα ερωτήματα. Επίσης η ψηφιοποίηση και, και ο ξεχρονισμός είναι φυσικά πολύ ενδιαφέροντα, όμως και η κυρία Νίμπλερ ήδη ανέφερε τις δικές της ε, ε, ανησυχίες τώρα για τις ε, νεοσύστατες εταιρείες να σας πω ότι το 97% των ε, μονοπρόσωπων εταιρείων αυτών είναι αυτοαπασχολούμενοι που είναι στην ουσία ψευδής αυτοαπασχόληση. Γι' αυτό λοιπόν συμπερασματικά μπορώ να πω ότι αυτή η πρόταση δεν είναι η πρόταση που θα δώσει λύσεις. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια έκκληση αντί της πρότασης αυτής να γίνει μια καινούργια πρόταση που θα αντιμετωπίζει αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ θα θέλατε να κάνετε μία σύντομη δήλωση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, εκτιμώ το γεγονό ότι μου δώσατε το λόγο. Ε, είμαι στην Επιτροπή ίνκο και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή ίνκο για το θέμα αυτό θα γίνει στις 29 Ιουνίου. Φυσικά και υπάρχουν συζητήσεις σε άλλες επιτροπές και στις πολιτικές ομάδες, όμως φρονώ ότι η πρόταση αυτή συνάδει απόλυτα με τις στρατηγικές προτεραιότητες τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσωπικά τη στηρίζω διότι πιστεύω πω θα δώσει όθηση στην ανταγωνιστικότητα, θα μειώσει το κόστο και θα δημιουργήσει ένα καλύτερο περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα. Παρά του συμβιβασμού που θα χρειαστεί να κάνουμε, πρέπει να κρατήσουμε την ουσία τη πρόταση αυτή, δηλαδή να δημιουργείται με χαμηλό κόστος και με μεγάλη ταχύτητα ηλεκτρονικά μια νέα εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να δρομολογηθεί και η ψηφιοποίηση της ενιαίας αγοράς. Αυτή είναι η προτεραιότητα του θέματος αυτού. Και πώς έχουν τα πράγματα σήμερα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν τα δύο τρίτα των ε, θέσεων απασχόλησης. Υπάρχει όμως, υπάρχουν όμως πολλές δυσκολίες στην ε, διασυνοριακή δραστηριότητά τους. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως η πρόταση αυτή είναι η καλύτερη που μπορούμε να έχουμε για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πασκόλου Τεγκράντες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ε, για την υπομονή σας. Νομίζω ότι η επιφυλακτικότητά μου ήταν απόλυτα αιτιολογημένη. Ευχαριστώ αυτά που μας είπε η Προεδρία που έκανε θαυμάσια εργασία και ευχαριστώ και τη θετική διάθεση της νέας Προεδρίας που θέλει να συνεχίσει να ασχολείται με το θέμα αυτό αλλά ακούσαμε και διάφορους βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, πολύ έντονες και διαφορετικές απόψεις. Γι' αυτό προτείνω πρέπει να κάνουμε μια συνεδρίαση των ε, σκιωδών στο Στρασβούργο για να ακούσουμε και λαμβάνω υπόψη αυτά που είπε ο κύριος Βος ότι θα μπορούσαμε να βρούμε και ένα άλλο τριμερή ανεπίσημο διάλογο για να δούμε κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει αυτό το θέμα. Θα προσπαθήσουμε ε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το να πάμε πολύ γρήγορα δεν έχει έννοια. Εγώ πρέπει να καθορίσω το χρονοδιάγραμμα για να δούμε τι μπορεί να γίνει και δεν μπορεί να γίνει. Και θα σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα αυτών των περαιτέρω συζητήσεων και να δούμε αν θα είναι ε, επικοδομητική όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Το 24 της κυρίας Κάουφμαν θα συζητηθεί το απόγευμα. Ευχαριστούμε τους Γερμηνείς για την υπομονή τους. Ευχαριστώ για την συμμετοχή σας.